Uh, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω αμέσως από το πρώτο σημείο της ημέρας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης υιοθετείται ως έχει ανακοινώσεις. Να σας ανακοινώσω ότι έχουμε διερμηνία διαθέσιμη σε 18 γλώσσες και η συνεδρίαση μεταδίδεται και ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Έχουμε συστάσει των συντονιστών, να σας πω σε αυτό, έχουν διανεμηθεί ηλεκτρονικώς, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται ως εγκεκριμένες προτάσεις. Πάμε τώρα στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το πραγματικό του ουσιαστικό θέμα. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον κύριο Λοράν Φαμπιού, στην Επιτροπή περιβάλλοντο για ανταλλαγή απόψεων για την προετοιμασία για την COP21 για τη διάσκεψη την αλλαγή του κλίματος που θα λάβει χώρα στο Παρίσι το Δεκέμβριο. Πέρα το ότι είναι υπουργό εξωτερικό της Γαλλίας, ο κύριος Φαμπίου είναι πρόεδρος της COP21 και θα έχει κρίσιμο ρόλο στην προεδρία της συνεδριάσεως που έχει μεγάλη παγκόσμια σημασία βλέπουμε στο να ακούσουμε ποιε είναι οι απόψει ενός Υπουργού αντιπροετοιμασία τη προετοιμασία της κυρίως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας ad hoc για την πλατφόρμα του Durban για την ε, δράση για τις αλλαγέ ε, και έγιναν ε, διάφορες διαπραγματεύσει στη Βόνη από αυτού. Θέλουμε να ξέρουμε τι περιμένετε από τη διάσκεψη όσον αφορά μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο για, την, για το κλίμα και έχουν υποβληθεί κάποιες προτάσεις ε, και τι μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση ενέργεια του κλίματο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα στείλει 15 μελή επιτροπή στη διάσκεψη και θα έχω την τιμή να προεδρεύω τη αντιπροσωπεία εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη αντιπροσωπεία αυτού. Κατανοούμε τη σημασία που έχει να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλεί με μία φωνή κατά τη διάρκεια τη διασκέψεω. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε παντιοτρόπω για να επηρεάσουμε τι διαπραγματεύσει θετικά. Ε, σήμερα χαιρόμαστε που έχουμε και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόκ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έλμαρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να προβώ σε κάποια σχόλια. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος που ασχολείται με το θέμα αυτό Έχουμε υποβάλει τη γνωμοδότησή μας για τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων το Δεκέμβριο. Η παρούσα κατάσταση με το κύμα αυτό των προσφύγων που αντιμετωπίζουμε ε, δεν έχει κορυφωθεί και αυτό σχετίζεται το πρόβλημα με την αλλαγή του κλίματος, αλλαγή του κλίματος, νερό, όλα αυτά τα, θέματα ε, γίνονται όλο και πιο σημαντικά θέματα γεωπολιτικά και όχι αποκλειστικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Ε, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προοπτικέ των λαών που ζουν εκεί. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τι συνθήκε, θα πρέπει να εξετάσουμε και την αλλαγή του, του κλίματο. Στην Επιτροπή λοιπόν των Εξωτερικών ε, Υποθέσεων, θέλουμε να ενθαρρύνουμε, σαν Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντο να αναγνωρίσει τη σχέση που υπάρχει ε, και να καταφέρουμε να ακολουθήσουμε μια επιτυχή πολιτική και να είναι επιτυχή η διαπραγματεύση στο Παρίσι. Ήδη συνομίλησα με τον Υπουργό επ' αυτού και είμαι πεπισμένος μετά από τη συνομιλία μας ότι αυτή η διασύνδεση μεταξύ μετανάστευσης, ειρήνης και πολιτικής για το κλίμα ε, είναι πολύ στενή ε, και είναι απαραίτητο να εξεταστεί αυτό και να εξεταστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, αντιμετώπιση να αναπτύξουμε μια στρατηγική, μια πολιτική σχετική. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό και την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη δυνατότητα της συνεργασίας που μας παρέχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλμαρ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λεωράν Φαμπιούς για να προβεί στα εισαγωγικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους παραόντες και όλες τις παρούσες. Είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να παίρνω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μιλήσω για τη διάσκεψη των μερών 21 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι και την οποία θα έχω την τιμή να προεδρεύσω και στην οποία θα έχω την τιμή να προεδρεύσω. Δεν θα ήθελα να κάνω μια γενική εισαγωγή, κάποιες γενικές ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Αντιθέτως, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα ε, να μιλήσω για το πώς ε, έχει η κατάσταση, κατά την άποψή μου, σήμερα τώρα. Δεν θα κάνω γενική, περιγραφή του, του θέματος, όμως θέμενη αξία πιστεύω ότι θα κομίσω εάν καταφέρω να σας ε, ε, εκφράσω την άποψή μου για την κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Στη... Είχαμε την διαπραγμάτευση της ομάδας NDP την περασμένη εβδομάδα. Ε, το κείμενο ήταν σύντομο, δεν έγινε δεκτό. Η διαπραγματεύση ήταν αρκετά έντονες δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα κείμενο με βάση το μέγεθός του, αλλά μετράει και το μέγεθος, περίπου περίκταση του κειμένου. Πάρα πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά. Από την άλλη να μην είμαστε ε, υπέρ της καταστροφολογίας. Ξέρετε, στην Κοπεχάγη το κείμενο είχε έκταση 200 σελίδων. 50 ε, σελίδες είναι καλύτερο από πλευράς έκτασης και μεγέθους κειμένου. Ωστόσο, πολλά σημεία παραμένουν ανοιχτά, παρόλο που έχουμε σημειώσει πρόοδος, να μην υπερβάλλουμε κιόλας στην ε, απεσιόδοξη πλευρά. Επομένως μέχρι τη διάσκεψη σε όλο αυτό το μήνα που θα μεσολαβήσει θα συνεχιστεί η δουλειά μας. Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στη Παρίσι θα έχουμε την pre-COP, την πρώτερη προκαταρκτική διάσκεψη των μερών με 80 περίπου υπουργούς για να συζητήσουμε θέματα επί της ουσίας και να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε σε βάθος. Δύο άτυπες συνεδριάσεις και συσκέψεις με αυτό το θέμα έχω ήδη οργανώσει και ήταν χρήσιμες και ελπίζω ότι ε, σε αυτή την ε, προκαταρκτική σύσκεψη εν ώψη της ΚΟΠ την επόμενη εβδομάδα με τους 80 υπουργούς θα σημειώσουμε πρόοδο ελπίζω. Έχουμε στη Μάλτα συνεδρίαση των χωρών της κοινοπολιτείας στην παραμονή της ΚΟΠ και έχουμε και το G20 στην Τουρκία. Είναι δύο σημαντικά ε, γεγονότα που παρεμβάλλονται μέχρι την ΚΟΠ του Δεκέμβρη στο Παρίσι. Και έχουμε και την Κίνα, θα μεταβώ στην Κίνα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα έχουμε εκεί συσκέψεις με τους Κινέζους ομολόγους μας και θα προβλέψουμε ε, ζώνες προσγείωσης, ε, σημεία στα οποία μπορεί να σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με τη θέση της Κίνας και την θέση της Γαλλίας αντιστοίχως. Με όλα αυτά θα φτάσουμε στις 30 ε, Νοεμβρίου, Η έναρξης της, έναρξης της διάσκεψης ε, των μερών. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα παρέμβουν την πρώτη μέρα. Αυτό είναι διαφορετικό και είναι και η καινοτομία. Στην Κοπεχάγη οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, είχε προβλεφθεί να συνεδριάσουν στο τέλος γιατί είχαμε σκεφτεί ότι ε, θα μπορούσαν ε, στο τέλος να λύσουν τα ε, τα ζητήματα. Εμείς αλλάξαμε γιατί δεν μπορεί σε ένα βράδυ να λυθούν όλα και θεωρήσαμε ότι οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να έρθουν στην αρχή ακριβώς για να στείλουν το ισχυρό πολιτικό μήνυμα και στη συνέχεια εμείς να κάνουμε την τεχνική δουλειά. Γι' αυτό και απευθύναμε πρόσκληση για την πρώτη μέρα, την παρουσία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων την πρώτη μέρα και ήδη 80 μας απάντησαν καταφατικά. Στη συνέχεια έχουμε το κείμενο της Βόνης, η τεχνική δουλειά θα γίνει πάνω σε αυτό. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας αυτό το κείμενο έτσι όπω θα έχει προτροποποιηθεί μέχρι τότε θα έρθει στα χέρια των Υπουργών και θα προσπαθήσουμε να το δέσουμε, να το ολοκληρώσουμε εκεί. Εγώ είμαι εδώ ως εκπρόσωπος και πρόεδρος της ΚΟΠΤΕ, τη διάσκεψης των μερών ε, για το κλίμα, για την κλιματική κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 21 στο Παρίσι και όχι ως εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης σήμερα. Ε, έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και θέλουμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό, να συμφωνήσουν όλοι επί του κειμένου για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξουν και συμβιβασμοί όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, επί της ουσίας, αυτά ως ε, γενικότερο πλαίσιο και διαδικαστικό. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας, τι θα σημαίνει μια επιτυχία της διάσκεψης των Παρισίων 21 ε, για την κλιματική αλλαγή πώς θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει επιτυχία. Πρώτον, εάν υπάρχει συμφωνία, εάν καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία νομικώς δεσμευτική, η οποία θα επιτρέψει να περιοριστεί πράγματι αποτελεσματικά η η κλιματική θέρμαση του πλανήτου κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου στα επόμενα 10 ε, με 20 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο ε, θα μας ικανοποιήσει. Αν υπάρχει τέτοιου είδους νομικός δασμευτική συμφωνία που θα έχει τέτοιες προβλέψεις, αυτό σημαίνει ότι η διάσκεψη των μερών και η διάσκεψη των Παρισίων θα είναι επιτυχημένη. Θα έχει στεφθεί με επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση ε, βλέποντας τις δεσμεύσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ μπορώ να διαπιστώσω ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πάνω μέρος της κλίμακας αυτής. Πέρα από τη φιλόδοξη αυτή ε, συμφωνία θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τι έχει γίνει ε, τα τελευ... τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με το ENDC, τις συνεισφορές δηλαδή. 154 χώρες έχουν καταθέσει τις συνεισφορές τους σε σχέση με το 90% των εκπομπών ενώ το ποσοστό 15% στο παρελθόν. Δεν θα ήθελα προς το παρόν να ταξινομήσω τις συνεισφορές, ε, τη συμβολή της κάθε χώρας, αυτό που έχει καταθέσει δηλαδή ως πρόταση για να μειώσει, όμως γιατί διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη, όμως είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός ότι 154 χώρες που που τελικά θα φτάσουμε στις 180 θεωρώ και ελπίζω. Έκαναν το διάβημα να αναρωτηθούν ως χώρες ποια πρέπει να είναι η πολιτική μας, η ενεργειακή, η πολιτική μεταφορών για τα επόμενα χρόνια και πώς θα συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών κτλ. Το γεγονός ότι αναρωτήθηκαν 154 χώρες αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Έχουν άλλωστε προθεσμία μέχρι την 1η Νοεμβρίου να καταθέσουν και οι υπόλοιπε χώρε τη συνεισφορά του και η Γραμματεία ε, θα αποφανθεί την 1η Νοεμβρίου. Ήδη όμω έχουμε κάποιε αξιολογήσει. Τι λένε οι εμπειρογνώμονε. Εάν δεν κάνουμε τίποτα θα πάμε σε 4, 5 ή 6 βαθμούς ε, παραπάνω θερμοκρασία. Δική μας φιλοδοξία είναι να φτάσουμε στο συν 1, 2 μόνο. σύμφωνα με τη γραμματεία ίσως μπορεί να κινηθεί όλο αυτό το πράγμα γύρω στο 2,7 με 3. 2,7 με βαθμούς. Είναι αρκετά καλά, είναι πολύ καλύτερα και σίγουρα πρέπει να γίνει παραπάνω δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα κριτήρια της επιτυχίας ε, θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή η έξτρα δουλειά. Η ρήτρα αναθεώρησης είναι το στοιχείο κλειδί και βεβαίως εγώ πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Εάν κάτι όμως πρέπει, για κάτι πρέπει να αγωνιστώ είναι το εξή. Στη Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να μπει ένας μηχανισμός αναθεώρησης. Όλο και πιο πολλές αντιπροσωπείες λένε ότι θα πρέπει να γίνεται κάθε πέντε χρόνια, ο οποίο μηχανισμός θα μας επιτρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε, να δούμε τη συνεισφορά της κάθε χώρας, τη συμβολή της σε αυτόν τον αγώνα. Εάν καταφέρουμε να ε, έχουμε ε, αυτά τα δύο σημεία στο κείμενο, πρώτον συμφωνία, δεύτερον νομικός δυσμευτική, τρίτον μηχανισμό αναθεώρησης που θα μας επιτύχει τους τεχνικούς μας στόχους, θα είναι τότε η διάσκεψη των Παρισίων, αυτό το οποίο σε άπτες στο γαλλική αποκαλούμε turning point, σημείο καμπής δηλαδή. Και θα είναι καθοριστική. Ένα, μια άλλη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι να είναι, όπως σας είπα, νομικώς δεσμευτική η συμφωνία. Δεν θα σας μιλήσω για τις λεπτομέρειες του πώς ορίζεται ε, στο δίκαιο η νομικώς δεσμευτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει και η κοινή γνώμη και τα κράτη-μέλη και τα κράτη αυτά αυτά να έχουν τη βεβαιότητα ότι δεν είναι μια γενική πολιτική συζήτηση, είναι μια συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπουν φυλακοί όσοι δεν την εφαρμόσουν, αλλά ότι υπάρχει μια νομική συγκεκριμένη μετάφραση αυτής της συμφωνίας, Και είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση. Τώρα, νομικός δεσμευτική θα είναι μόνο για τις πλούσιες χώρες ή και για τις χώρες που δεν έχουν τη φήμη ότι είναι πλούσιες θα ήταν ευκταίο και επιθυμητό αυτό να αφορά τους πάντες παρόλο που υπάρχουν δύο βαθμοί δέσμευσης. Τρίτη προϋπόθεση επιτυχίας είναι η χρηματοδοτική και τεχνική τεχνολογική πλευρά. Όταν συζητάει κανείς με διάφορες αφρικανικές χώρες μας λέ, ακούει ότι κοιτάξτε έχετε δίκιο αλλά εμείς δεν ευθυνόμαστε για τα αέρια ε, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ε, και είμαστε και μάλιστα θύματα αυτής της κατάστασης και θέλουμε τεχνολογία και χρηματοδότηση. Και ακούγεται αυτό λογικό. Και σύμφωνα με τη μελέτη του ΩΣΑ γνωρίζουμε ότι το 2014 θα φτάσουμε, έχουμε προχωρήσει στο στόχο των 100 ε, δισεκατομμύριων και θα, θα προχωρήσουμε και θα το ξεπεράσουμε κιόλα. Και αν καταφέρουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα στο Παρίσι, τότε πιστεύω ότι θα είναι μία επιτυχημένη ε, διάσκεψη. 11 λεπτά και 24 ε, δευτερόλεπτα. 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα ξεπέρασα το χρόνο μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ξεκινώντας με τον τονιστές. Πίτερ Λίζε για το ΕΛΚ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Τζοβάνι. Χαίρομαι πραγματικά που με τις δύο κοινοβουλευτικές μας επιτροπές από κοινού συνεδριάζομαι. Αυτό που είπε ο Έλμα Μπρόκ, ότι φυσικά οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και το πεντάγωνο στη ΣΥΠΑ μεταξύ το δημοσιοποίησε αυτό. Και έχουμε και μια διπλωματία για το κλίμα και στην εξωτερική μας πολιτική στις προσπάθειές μας προσπαθούμε οι στόχοι για το κλίμα, για τη διεθνή πολιτική πάντα να συμμετέχουν όταν διαπραγματεύομαστε με τρίτες χώρες. Κύριε Υπουργέ, δίκαια και σωστά είπατε ότι μέχρι σήμερα δεσμεύσεις των κρατών μελών δεν επαρκούν ώστε ο στόχος αναχέτησης σε δύο βαθμούς της υπερθέρμανσης του πλανήτη για μην μιλήσουμε για λιγότερο το 2% πρέπει να έχουμε υπόψη στόχο και φυσικά πολλή δουλειά πρέπει να γίνει αλλά είναι μια ιστορική ευκαιρία και το είπατε και αυτό 154 χώρες που ήδη τα στοιχεία τους τα έχουν δώσει και τεκμηριωμένα και γι' αυτό είναι αποφασιστική σημασία να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε αυτή τη διαδικασία να μην δημιουργηθεί στο Παρίσι μια κατάσταση αυτή η κατάσταση που είχε στεφθεί με επιτυχία να υπονομευθεί να χάσει το κύρος της ή να διακοπεί θέλω να σας ενθαρρύνω λοιπόν και θέλω την προσοχή σας να τη στρέψω σε ένα ιδιαίτερο τομέα <clears throat> στις ε, διεθνείς ε, εναρίες μεταφορές. Ε, έχουμε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για τις εκπομπές τρύπων όσον αφορά τη βιομηχανία και κατά 43% όλα και πολλές βιομηχανίες ιδιαίτερα η χαλιβουργία πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Όμως έχουμε μηδενικό, μηδενικό επαναλαμβάνω επίπεδο στις εκπομπές ρήπων από τις αερομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές δεν υπάρχει ούτε αυτό. Λοιπόν πρέπει να υπάρξει σαφή εντολή προς τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εναέριες μεταφορές να συμμετάσχουν και να δεσμευθούν. Δεν μπορεί να εξαιρούνται αυτές, ενώ οι άλλες δεσμεύονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ζιλ Παγνιό, για τους σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ, κυρία Υπουργέ, εδώ στι επιτροπέ μα, στι κοινοβουλευτικέ συζητάμε την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο και πάνω σε αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ευρωκοινοβούλιο για να βοηθήσει στην επιτυχία τη Συνόδου Κορυφή των Παρισίων. Διευκολύνει λοιπόν την υλοποίηση τη διεθνού τη συμφωνία για το κλίμα. Και ε, έχουμε φιλοδοξία να είναι επιτυχή αυτή η διάσκεψη. Και το αναφέρουμε και στην έκθεση τη οποία έχω την τιμή να είμαι εισηγητή, όπω αναφέρατε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να χαιρετήσω επίσης τη δέσμευση την προσωπική που αναλάβατε για την επιτυχία της συμφωνίας. Η παρουσία σας στη Βόνη εξάλλου αρχές της περασμένης επέτρεψε μια νέα όθηση πολιτική να δοθεί στι διαπραγματεύσει μερικέ εβδομάδε πριν να αρχίσει η ΚΟΠ στο Παρίσι έναντι των αυξανωμένων ησυχιών ε, των χωρών του G77 ε, και αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Μετά από τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, όπως υπενθυμίσατε κύριε Υπουργέ, στην Βόνη έχουμε πιο μακροσκελές κείμενο, αλλά καθορίζονται διάφορες επιλογές και δυνατότητες για να επιτευχθεί συμφωνία στο Παρίσι και έτσι μέσα στις λύσεις να βρούμε διέξοδο. Και στο, στην έκθεσή μας του Κοινοβουλίου αναφέρουμε κάποια σημεία που είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για την COP21. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι τα 100 δις ευρώ το χρόνο μέχρι το τέλο του 2020, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε έναν οδικό χάρτη ευρωπαϊκό που θα καθορίζει πώ δεσμεύεται ο καθένα κάθε κάτω μέρος, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτό το ταμείο, το πράσινο. Μετά καινοτόμω χρηματοδότηση, το ταμείο, το πράσινο αυτό, δεν μπορεί μόνο του να καλύψει την όλη μετάβαση προ μια οικονομία που δεν θα εκπέμπει άνθρακα, δεν χρησιμοποιεί άνθρακα, να αλλάξουμε νοοτροπία οικονομική να σταματήσουν οι επιδοτήσεις για τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ε, το είπαμε, είναι επίση πολύ σημαντικό να το επενθυμίσουμε. Και τέταρτον, να όλοι οι φορείς να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στην έκθεσή μας. Έχουμε υπογραμμίσει τη σημασία που έχει το θεματολόγιο με τις λύσεις. Ιδού εν ολίγης, εντός διλέπτου, ε, τι ήθελα να σας πω και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε παρόντες υπό την προεδρία του κ. Λαβία στην αντιπροσωπεία την επίσημη του Ευρωκοινοβουλίου, στην ΚΟΠ, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να επιτύχει αυτή η σύνοδος. Julie Gerling για το ECR, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Φαμπιούς. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα αφορά τις προθέσεις σας που θα έχετε ως πρόεδρος στην ΚΟΠ. Πώς θα προβείτε στις διάφορες δημόσιες ανακοινώσεις σας στις βιομηχανικές χώρες που αφορά αυτό όλη την Ευρώπη υπεκρατεί ε, μια κάποια ανυπομονησία άρχισε ανυπομονησία όσον αφορά αυτή την συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο διότι κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες αλλά και αλλού ότι κλείνει η χαλιβουργία μας διότι παράγεται ο χάλιβας αλλού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος και έρχεται στην αγορά το προϊόν αυτό και σε περιπτώσεις συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου πρέπει να κάνουμε κάτι για το dumping αλλά είναι δύσκολο. Και χάνει την υπομονή του το κοινό διότι ακούγονται κλήσει να ξοδεύονται μεγάλα ποσά, 100 δισεκατομμύρια ευρώ που το λένε πολύ εύκολα οι πολιτικοί, ε, το αναφέρουν το ποσό, αλλά δεν έχουν ακούσει τίποτα τι θα γίνει με τι θέσει απασχόλησή του, με τη δουλειά του. Και ε, χάνουν την υπομονή τους. Όλοι λένε τελικά όλα θα πάνε καλά στο τέλος των συνομιλιών και θα σωθεί ε, η γη, θα καταπολυθεί η αλλαγή του κλίματος και αυτό δεν είναι αληθές. Εάν έβλεπε ο κόσμος ότι ε, αναλαμβάνεται συγκεκριμένη δράση αλλού θα συμφωνούσαν. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη στην COP21 να γίνει κάτι, να δώσει αποτελέσματα, να φανεί ότι αναλαμβάνονται δεσμεύσεις από τον υπόλοιπο κόσμο να κάνουν κάτι και οι άλλοι. Και αντί να γίνονται τέτοιες δηλώσεις μεγαλόσχημες και να κατηγορούνται κάποιοι και να λέμε ότι εμείς πρέπει να γηθούμε για να αλλάξουμε το κλίμα θα πρέπει κάποιος άλλος τρόπος να υπάρξει να διαβιβαστεί σωστά το μήνυμα και το ερώτημά μου είναι αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το δώσετε αυτό το μήνυμα αυτόν τον τρόπο ευχαριστώ ο κ. Γκερμπράντι από την ΑΝΤΕ ευχαριστώ Πρόεδρε Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Φαμπιούς για τα αρχικά σας ε, σχόλια. Θα επικεντρωθώ επί κάποιες προτεραιότητα σας, δηλαδή τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των του κλίματος. Σας συγχαρώ τη Γαλλία, διότι έχει ηγηθεί στις προσπάθειες στον τομέα και έχει ε, προσημειώσει και δεσμεύσει ε, δισεκατομμύρια για την καταπολέμηση του φαινομένου. Έχω κάποια ανησυχία όμως. Ποια θα είναι η χρηματοδότηση για το θέμα αυτό μετά το 2020. Οπότε εδώ μπαίνει και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολό της, τι ρόλο θα παίξει. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι πολλές χώρες που θα είναι στην COP21 έχουν θέσει αυτό σαν κριτήριο, σαν κριτήριο. Μπορούν να συμφωνήσουν επί φιλοδόξου κειμένου τη ΣΚΟΠ αν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση. Στι 10 Νοεμβρίου έχουμε συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Κρισίμου σημασία για την ευρωπαϊκή θέση. Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που συντάχθηκε από τον Ζιλ Παγνιού ζητήσαμε στο ETS να μπουν στο αποθηματικό κάποια ποσά μετά το 2020 για να υπάρξει επαρκής ε, κάλυψη χρηματοδοτική από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έχετε να πείτε κάτι όσον αφορά το επικείμενο, ε, την επικείμενη σύνοδο του ΕΚΟΦΗΝ και ποιε δεσμεύσει πιστεύετε θα αναλάβει η χρηματοδοτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για μετά το 2020. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο κ. Σομαρή για την Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση γενικής φύσεως και να θέσω και συγκεκριμένη ερώτηση. Βλέποντας λοιπόν τις συνδυασμένα αποτελέσματα της αύξησης του πληθυσμού στον κόσμο, της συνέχισεως του οικονομικού μοντέλου που έχει ξεπεραστεί να εφαρμόζεται και τη διάδοση τρόπων ζωής που βασίζεται στα πρότυπα τα αμερικανικά ή ευρωπαϊκά Όλα αυτά δείχνουν τη δυσκολία που έχετε μπροστά σας για να συγκρατήσετε τη θέρμανση του πλανήτη και να παραμείνει κάτω η θέρμανση αυξής θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς και πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον παράγοντα χρόνο. Δεν είναι πολύ αργά αλλά ήδη είναι αργά. Γίνονται διασκέψεις η μία μετά την άλλη οι οποίες περιπλέκουν την υλοποίηση ε, και την επίτευξη του στόχου. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω αφορά τα νησιά. Βλέποντας ένα χάρτη του κόσμου, βλέπουμε από τη Μεγάλη Αυστραλία μέχρι τις μικρές ατόλες έχουμε 300.000 ε, νησιά και παίζουν ε, ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο προσκήνιο το παγκόσμιο εν ώψη της αλλαγής του κλίματος. Βλέπουμε πόσο μικρές χώρες όπως το Κυριμπάτι ε, σήμερα ε, είναι στο προσκήνιο το παγκόσμιο. Λοιπόν, και μεταξύ των 300.000 νησιών υπάρχουν ευρωπαϊκά νησιά που αντιμετωπίζουν την, είναι πιο εξίσου ευάλωτα όπως τα μικρά νησιά, τα μικρά νησιωτικά κράτη που αναπτύσσονται. Και ανάμεσα στα ευρωπαϊκά νησιά υπάρχουν οι υπερπόντιες ευρωπαϊκές νήσοι, υπερπεριφερειακές νήσοι ε, και υπερπόντια εδάφη και επικράτης. Και έχουμε το συνέστημα ότι αυτά τα μικρά ευρωπαϊκά νησιά έχουν μείνει στο περιθώριο των ισχυρών δικτύων που δημιουργήθηκαν από τα μικρά ε, νησιά τα άλλα ε, και δεν υπερασπίζονται σωστά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών νησιών όσον αφορά την προσαρμογή στο κλίμα. Ε, λοιπόν, Ποιους μηχανισμούς προβλέπετε, ποιες λύσεις προβλέπετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα όσον αφορά αυτά τα ευάλωτα ευρωπαϊκά ε, νησιά. Ευχαριστώ. Ο κ. Σαγέντο για τους Πρασίνους. Κύριε Υπουργέ καλημέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ, είναι σημαντικό. Ε, εάν είναι επιτυχή η διάσκεψη αυτή, θα είναι επιτυχία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και δική σα. Και αν είναι αποτυχία, θα είναι αποτυχία του ΟΗΕ. Αλλά είναι σημαντικό να είσαστε παρόντες. Ε, διότι κατά βάθο αυτό δεν αρκεί βέβαια, αλλά θα υπάρχει επιτυχία αν δεν υπάρχει ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις διαπραγματεύσεις. Και σας ευχαριστώ που ηγείστε των προσπαθειών. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Ζεμπράντη, θέλω να σταθώ στη χρηματοδότηση. Στις 14 Νοεμβρίου ελπίζουμε ότι στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ θα υπάρξει και μια συμφωνία όσον αφορά την φορολόγηση των χρηματοστικών συναλλαγών. Στο πεδίο εφαρμογής δηλαδή ε, ξέρουμε την αρχή και τις λεπτομέρειες. Ε, ουσιαστικά πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει και για το G, για G20 και για την COP21 να καταλήξει με μια ανακοίνωση 11 χώρε Ευρωπαϊκή Ενώσεω που μπορούν να προβούν σε μια ανακοίνωση επί του θέματο χρηματοδοτήσεω που θα είναι σαφέστερη σε σχέση με, την, ε, με τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα μπορέσει να ανακοινωθεί κάτι εκεί. Και α μην είναι άμεσα θέμα τη COP21. Τέλο, δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει δεσμευτική α, ε, συμφωνία στον αφορά τι υποχρεώσει με επιβολή κυρώσεων ε, λοιπόν, η αξιοπιστία επίσης των δεσμεύσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το σύστημα του ελέγχου, της επαλήθευσης που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί αξιοπιστία σε όλα αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό διότι είδαμε ακόμα και χτες ότι έχουμε ένα σαφή στόχο που είναι η οδηγία 2 ε, και 5 και 6 για τις ε, ε, εξατμίσεις των αυτοκινήτων που συμφωνήθηκε το 2007 και παρόλα αυτά είπαν ότι παράλληλη τη συμφωνία μπορεί να διπλασιάσουμε τη μόλιση κατά, επί σειρά ετών. Άρα τελικά αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία των μέτρων που λαμβάνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η FTD, ο κύριος Έλμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Ιδιαίτερα με εξέπληξε, εντυπωσιάστηκα την ελπίδα σας ότι θα περιορίσουμε σε 2,73 βαθμούς ε, την υπερθέρμανση του πλανήτη η ιστορία της ε, ιστορίας καταπολέμησης των αλλαγών του κλίματος ε, είναι ότι πολλές φορές έχουν πέσει έξω οι προγνώσεις και αυτό το ότι εσείς κάνετε τώρα προβλέπετε με μάλιστα κατά ένα εκατοστό βαθμού ε, Κελσίου την τροχοπέδηση της υπερθέρμανσης παρα, καταλήγει σε κάτι παράλογο καταλήγουμε στην διάσκεψη των Παρισίων και ψάχνουμε να βρούμε μια δεσμευτική συμφωνία είναι ο θρίαμβος της ελπίδας ε, επάνω στην πύρα Κάθε φορά ελπίζουμε θα τα καταφέρουμε και αποτυγχάνουμε. Κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ρόλο πρωτοπόρου, κανεί δεν ακολουθεί όμω. Το αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη υπονομεύει την οικονομία μα. Έχουμε ενεργοβόρε εταιρείε που τι διώχνουμε από την Ευρώπη. Χαλιβουργία. Η κυρία Γκέρλινγκ μίλησε για τα προβλήματα τη χαλιβουργία. Αλλά τα ίδια ισχύουν και για τη χημική βιομηχανία, και πολλές εταιρείες ε, εξωθούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε σε χώρες με χαμηλότερες ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, π.χ. Κίνα το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν ότι οι πραγματικές ε, εκπομπές λοιπόν θα αυξηθούν διότι οι ενεργοβόρες ε, εταιρείε ε, διώχνονται από την Ευρώπη και πάνε αλλού όπου οι προδιαγραφές είναι χαμηλότερες. Λοιπόν, πολιτική, ενεργειακή, <clears throat> κλιματική που δημιουργεί απίστευτη ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι παγκόσμιες εκπομπές ρήπων. Πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο παράλογος κύκλος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντονάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που είστε παρόν. Ευχαριστώ που μα δίνετε την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων σε ένα τόσο σοβαρό και δυσεπίλητο πρόβλημα. Δεν νομίζω θα αντιμετωπίσουμε τις δύο βασικές δυσκολίες όπως η πολιτική που θα σκηθεί στα πλαίσια του Πρασίνου Ταμείου θα υπάρξουν δράσει στο περιθώριο ίσως που θα μπορούσαν να διορθώσουν τις λειτουργίε όσον αφορά τους κανονισμούς και τι διατάξει των περιβάλλων και τα ανθρώπινα σφάλματα. Θα έχουμε παγκόσμιου στόχου, αλλά τελικά θα χειριστούμε τη ρήπανση και δεν θα αλλάξουμε πολύ το σύστημα που προφανώς καταστρέφει τον πλανήτη. Επίσης, και τη ρύθμιση ε, της που γίνονται για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές τι σχέδιο έχετε για να σταματήσουν εξάρτηση από τους ε, ε, ε, υδρογονάνθρακες κυρίως από τις, που προέρχονται από τις χώρες που είναι κυρίως ρηπαντές. Πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Νομίζω ότι τελικά αυτά τα θέματα βασικά δεν αντιμετωπίζονται και θα έχουμε περιορισμένα αποτελέσματα. Άλλη δυσκολία. Να, οι αναδυόμενες οικονομίες θα συμμετάσχουν στη συμφωνία. Αυτό είναι απαραίτητο για δύο λόγους. Αυτές οι χώρες αναπτύσσονται τώρα. Πρέπει να του δώσουμε κίνητρα να προβούν σαν αναπτύξη που είναι βιώσιμη και καθαρή. Οι χώρες οι αναπτυσσόμενες, κυρίως στην Ασία, ρηπαίνουν πολύ και ε, ρηπαίνουν περισσότερο από τα ευρωπαϊκά κράτη. Εφόσον από τι έμενε χώρε παραμένουν διστακτικέ όσον αφορά τι υποχρεώσει που αναλαμβάνονται για την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο, οι μόνε χώρε που μπορούν να κάνουν παραπάνω προσπάθειε θα είναι οι χώρε οι οποίε ήδη ασχολούνται πολύ με το κλίμα, όπω είναι οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Παρά τι προσπάθειε, οι προσπάθειές μας έχουν λιγότερη σημασία στο παγκόσμιο, ε, παγκόσμια κλίμακα και μειώνεται και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Δεν ομολόγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η μείωση των εκπομπών των αερίου του θερμοκηπίου στην Ευρώπη οφείλονται και στην οικονομική ε, ύφεση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και ότι η Γαλλία ε, ιδιαίτερο που εκπροσωπείται δεν θα έχει να δαπανίσει τόση ενέργεια για τίποτα, χωρίς να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Λοράν Φαμπιού, για να δώσει μία απάντηση, πρώτη ομάδα απαντήσεων στι ερωτήσει που ετέθεσαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους και όλες που μου έθεσαν ερώτηση αλλά και όσους και όσες δεν μου έθεσαν ερώτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μέσα σε 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου αλλά μην εκπλαγείτε βεβαίως εάν δεν απαντήσω ε, τόσο συγκεκριμένα όσο θα θέλατε. Ακούγοντά σας κράτησα κάποιες ε, σημειώσεις και παρατηρώ τώρα ότι ε, προκύπτουν συνεχώς ε, ορισμένα ζητήματα και θα ασχοληθώ με το πρώτο. Είπε κάποιος ότι αυτή η διάσκεψη είναι για το περιβάλλον αλλά όχι μόνο για το περιβάλλον και συμφωνώ απολύτως. Όλο και περισσότεροι πολίτες σε όλο τον πλανήτη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι απορριθμίζεται το κλίμα. Η δυσκολία έγκυται στο να τους καθησυχάσουμε, να αποδείξουμε τις δραματικές συνέπειες της μη δράσης, γιατί κόστος έχει και η δράση αλλά και η μη δράση, η αδράνεια και ε, άλλο, άλλη πρόκληση είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν εφικτές λύσεις Εάν περιγράψουμε τα πράγματα με εξαιρετικά δραματικό τρόπο χωρίς να ε, παρουσιάζουμε και λύσεις δεν θα πείσουμε κανέναν, ούτε θα λύσουμε και κάποιο πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό στη διάσκεψη, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο κλιματικό αυτό αυτό που είναι βέβαια, αλλά ότι αυτό το θέμα έχει εγκάρσιες συνέπειες, συνέπειες που διαπερνούν όλους τους τομείς μια κοινωνίας. Μιλούμε για τη σύντηση ή για το λοιμό, μιλούμε για την πλημμύρα ή για το, ε, τα βιώσιμα εδάφη. Μιλούμε για τον τρόπο ζωής ή για την μετανάστευση. Το κλίμα επηρεάζει όλους αυτούς τους τομείς. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για ε, πολλούς λόγους. Φανταστείτε ε, εάν πρέπει σε αυτούς να προσθεθούν και άλλοι για λόγους κλίματος. Είστε το θέμα του πολέμου, είστε το θέμα της ασφάλειας επίσης. Ε, επομένως ε, το δεν είναι αμυγός περιβαλλοντικό θέμα αλλά πολυσχηδές με πάρα πολλές προεκτάσεις. Επιπροσθέτως θα ήθελα να πω ότι δεν μίλησα αρκετά ούτε εγώ αλλά ούτε και εσείς για τους καθοριστικούς παράγοντες σε αυτή τη διάσκεψη οι οποίοι για πρώτη φορά θα είναι οι μη κυβερνητικοί εμπλεκόμενοι. Ο προκάτοχός μου κύριος Περούβια αλλά και εγώ ο ίδιος μετά τη διάσκεψη της Λίμα ε, του Περού το 2014 αποφασίσαμε ότι εφ' εξής, σε όλες τις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή θα υπάρχει ένα μέρος αφιερωμένο στους μη κυβερνητικούς παράγοντες δηλαδή στις κοινότητες, στις περιφέρειες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Άλλωστε, αν δούμε ποιο εκπέμπει αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όχι οι κυβερνήσεις άμεσα, έμεσα διότι οι κυβερνήσεις αποτελούνται από ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις. Όμως, όταν παίρνονται αποφάσεις για τη χή ε, ε, περιφέρεια και τις μεταφορές ή τα ε, απορρίμματα και την ψη επιχείρηση για το ενεργειακό αποτύπωμα και την χρήση άνθρακα κτλ. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή σε ποιο επίπεδο έχουν επιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις και γι' αυτό θέλουμε εκπρόσωποι και αυτών των επιπέδων να παραστούν, να, να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. 100 δις δολάρια το χρόνο αποφασίστηκε στη Κανκούν να κινητοποιούνται κάθε χρόνο από τις χώρες του Βορρά προς τις χώρες του Νότου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά μέχρι τώρα, από την Κανκούν μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε λογιστική καταγραφή του που βρισκόμαστε και αυτό ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Ο έκανε μια δουλειά πολύ σημαντική, δημοσιεύθηκε στη Λίμα πριν από κάποιες μέρες και σύμφωνα με τη μελέτη αυτή το 2014 η συνεισφορά των χωρών του Βορρά ε, στις χώρες της του Νότου ήταν στα 62 δις και μέχρι το 2020 πρέπει να φτάσει στα 100 δις. Θεωρώ ότι είναι εφικτό, είναι αναγκαίο, είναι δυνατό πριν τη διάσκεψη των Παρισίων να δείξουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στα 100 δισεκατομμύρια πριν το 2020 ή μέχρι το 2020. Έρχομαι τώρα στο πράσινο ταμείο το οποίο δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των 100 δις. 100 δις είναι διμερή κονδύλια, πολυμερή και δημόσια και μεταξύ αυτών υπάρχει και το πράσινο ταμείο το οποίο θέλουμε να πρικοδοτήσουμε όλο και περισσότερο. Σήμερα η αρχική του κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στα 10 δις αλλά θέλουμε να αποκτήσει πολύ περισσότερα. Και θα ληφθεί η σχετική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε καινοτόμε μορφές χρηματοδότησης. Το Συμβουλίο ΕΚΟΦΗΝ, ε, Συμβουλίο Υπουργών ε, Οικονομίας και Οικονομικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι θα λάβει χώρα στις 10 του μήνα και θα τεθεί το θέμα του φόρου επί του χρηματιστηριακών συναλλαγών. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να πάρει αυτό πιο συγκεκριμένη μορφή. Ε, άκουσα την ημερομηνία της 1ης Πρώτου του 2017. Η Γαλλία σε ό,τι την αφορά μεγάλο μέρος του φόρου το, επί των χρηματιστηριακών ε, ε, εναλλαγών θα το, να, θα το αφιερώσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. θετικό είναι όλες οι χώρες να αποφασίσουν να κάνουν το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία, αλλά σε κάθε περίπτωση όπως και αν θέλει κανείς, έστω τουλάχιστον να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση της εξέβρεσης καινοτόμου χρηματοδότησης. Οι τελευταίες μελέτες ε, που διαθέτουμε βλέπουμε, ε, μας δείχνουν ότι 500 δις ε, είναι τα χρήματα που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Μας λείπουν άλλα 100. Δεν έχουμε εντολή στη διάσκεψη των Παρισίων βεβαίως να αποφασίσουμε όμως, εάν τελικά θέλουμε να πάμε προς μια ενέργεια που, ενέργεια που χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο άνθρακα θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο δρόμους. Δηλαδή καταρχάς να αποτιμήσουμε την ενέργεια που βασίζεται στον άνθρακα και μετά να αποτιμήσουμε την ενέργεια που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές για να δείξουμε πόσο πιο συμφέρουσα είναι η δεύτερη αντί της πρώτης. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Πρώτα να αποδείξουμε ότι είναι σύμφορο το πρώτο και στη συνέχεια να αποδείξουμε ότι είναι πολύ πιο συμφέρον το δεύτερο. Δύο παράλληλες διεργασίες λοιπόν ως προς αυτό. Παρόλο που ως διάσκεψη δεν έχουμε εντολή να αποφασίσουμε ότι θα φύγουμε από τον άνθρακα συγκεκριμένα με νομικός δεσμευτικό τρόπο. Από εκεί και πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη ε, που να μην μας φέρει σε μειονεκτική και μη ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τις άλλες χώρες. Πράγματι, πρέπει την προσπάθεια να την καταβάλουν μόνο ορισμένοι ή όλοι με γενικότερο τρόπο. Όντως είναι ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα, από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Συμφωνώ με σας. Στις εργασίες όμως που κάνουμε παρατηρούμε ότι παρά τις διαφοροποιήσεις για το χύψη παράρτημα 2, την ε, ε, τάδε ή την άλλη ε, παράγραφο ή το ένα ή το άλλο εδάφιο, όλο και περισσότερο διαισθανόμαστε ότι υπάρχει γενικότερη συνέστηση του ότι όλες οι χώρες πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια. προσπάθεια. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει ε, την ίδια προσπάθεια από το Μαλή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βόρειες χώρες, οι πιο πλούσιες χώρες σίγουρα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό είναι προφανές και αυτονόητο. Αλλά όλοι όμως πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια και το σημαντικό είναι να περάσει το μήνυμα λέγοντας ότι ναι η δράση στοιχίζει λιγότερο από την αδράνεια αλλά δράση δεν σημαίνει ότι θα θυσιαστούμε εμείς ως Ευρωπαίοι ως Ευρώπη ε, θα είναι θυσία για όλους τώρα έρχομαι στο θέμα των νησιών όχι μόνο πρέπει, ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τα νησιά γενικά και στο σύνολό τους αλλά και επί τούτου και επί ε, πιο συγκεκριμένων θεμάτων. Και υπάρχουν εργασίες που έχουν ε, προβλεφθεί ε, συνεδρίες ειδικέ για τα νησιά και εκεί θα συζητηθεί ο μετριασμός, η απάλυνση του φαινομένου, του αντίκτυπου που θα έχει στα νησιά και η προσαρμογή των δράσεων στις ανάγκες των νήσων. πάντοτε μιλούμε για μετριασμό και για προσαρμογή, είναι οι δύο λέξεις κλειδιά. αξιοπιστία επαλήθευση όλων αυτών είναι θέματα που, στα οποία αναφερθήκατε και συμφωνώ απολύτως. Δεν θα είναι, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, μια συμφωνία ε, που θα ε, ε, διέπεται από το ποινικό δίκαιο. Προφανώς. Όμως πρέπει να είναι νομικός δεσμευτική και ε, κάθε λέξη μετράει ε, εάν θα ήταν θα πρέπει ή θα έκανε ή θα μπορούσε ε, οι χρόνοι μετρούν η, κάθε, η παραμικρή λεπτομέρεια στη διατύπωση του κειμένου μετράει έτσι ώστε να γίνει σεβαστή και να υπάρξει και μηχανισμός αναθεώρησης. Άλλωστε έχουμε και τεχνολογικές εξελίξεις που θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα και για να μην σας κρύψω τίποτα και να πω τα πράγματα με το όνομά τους θα έχουμε σύντομα δορυφόρους που θα πηγαίνουν πάνω από κάθε χώρα και θα βλέπουν πόσες εκπομπές ε, ε, του αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου ε, εκπέμπονται από τη συγκεκριμένη χώρα και πέντε χρόνια μετά μπορεί κανείς να επαληθεύσει κατά πόσο πραγματικά η χώρα αυτή έκανε την προσπάθεια που της αναλογούσε. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον παράγοντα τον χρονικό, του χρόνου. Ξέρετε, δεν είναι μία διαπραγμάτευση όπως οι άλλες. Ε, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, εάν ε, δεν πετυχαίνουμε συμφωνία ε, φέτος, μπορούμε να συνεργαστούμε του χρόνου, κάποια άλλη φορά. Όμως, τα αέρια του θερμοκήπου οποίου δεν εξαφανίζονται την επόμενη χρονιά, παραμένουν για δεκαετίες αν όχι για αιώνες και κάθε χρόνος που περνάει είναι σε βάρος μας και αν περάσουμε ένα σημείο καμπής τότε μετά η κατάσταση θα είναι μη αντιστρέψιμη, θα είναι αναντιστρεπτή. Θα πρέπει να δράσουμε τώρα, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν ε, ε τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχει όφελος και κέρδος που μπορεί να βγει από αυτό και θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, αρκετά προσεκτικοί αλλά και αρκετά τολμηροί επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε το δεύτερο γύρο. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους. Έχουμε πάνω από 27 που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ένα λεπτό, αλλά ένα λεπτό παρακαλώ ο καθένας. Στο ένα λεπτό πρέπει να σταματάμε. Φρανσουάζ Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ Προέδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς ευχαριστώ που είσαστε εδώ ανάμεσά μας για να ανταλλάξουμε απόψεις για τη διεθνή αυτή η διάσκεψη είναι πολύ σημαντική. Έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία η οποία θα είναι χρησιμότατη. Θα επιτρέψει την ε, εξέβρεση μιας λύσης, να καταλήξει κάπου η διάσκεψη. Δεν θα είναι κάπου, θα, θα είναι η βάση για να καταπολεθεί η αλλαγή του κλίματος. Υποστηρίζω θερμά το θεματολόγιο των λύσεων που θα συμπεριληφθούν στην ε, συμφωνία, που θα πρέπει να στοχεύει στις νέες τεχνολογίες που πρέπει να υποστηριχθούν, οι νέες ε, τεχνολογίες ε, με χαμηλές εκπομπές άνθρακος, θα πρέπει να διευκολυνθεί η χρήση τους, η ανάπτυξή τους, η σύλληψη, η αποθήκευση του άνθρακα, θα πρέπει να κάνουμε στάθμιση των υπέρ και των κατά των λύσεων και η ψηφιακή επανάσταση οδηγεί σε νέες μεθόδους εργασίας. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να αναλύσετε περισσότερο για, την, για το προσύμφωνο. Ασχολήθηκε με τις εφαρμογές στην ιδιωτικό τομέα και τη χρήση νέας τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ματίας Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Συγχαρητήρια, έπαινο, γιατί τη δομή της διάσκεψης την αλλάξατε να είναι ευθύ εξ αρχή οι αρχηγοί παρόντε, να μην χάνουμε χρόνο. Ο ίδιος, η ίδια πίεση να ασκείται και έναντι σε, για τον κρατών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θέλω να αναφερθώ να αλλάξει η κοινωνία, να αλλάξει η νοοτροπία μας, η βιομηχανία σας. Ε, είχα συναντήσει στην γενέθλια πόλη σας. Ε, με εντυπωσίασε ότι είχατε μια ιδέα βιομηχανοποίησης ε, με την ιδέα της αποσύνδεσης από την εκπομπή ρήπων διοξιδίου του άνθρακα. Η σωστή προσέγγιση μπορεί να γίνει αυτό, αλλά χρειαζόμαστε κανόνες. Και ο συνάδελφος Λίζε το ανέφερε. Χρειαζόμαστε ένα έπαθλο ε, για τον άνθρακα. Ε, μια τιμή, με συγχωρείτε, ένα αντίτιμο για τον άνθρακα, ώστε να είναι ακριβή η εκπομπή ε, αερίων θερμοκηπίου. Αυτά τα δύο θέματα λοιπόν να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους και τότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά. Thank ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Δύο παρατηρήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα η χαλιβουργία μας βρίσκεται πηξηρού άκμης. Αρκετοί το ανέφεραν. Αντιμετωπίζουμε σημαντικότερες προκλήσεις από το outsourcing και με το dumping με χαμηλότερες προδιαγραφές από άλλες χώρες και σε σχέση με την εισήγηση για το σύστημα εκπομπών ρήπων, πώς θα μπορούσε να συνδεθεί ένα σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας που θα έδινε ευκαιρία να τα καταφέρουμε. Αν το καταφέρουμε, τότε μπορούμε να ε, οδηγήσουμε και άλλες χώρες να ε, θεσπίσουν αυτές τις προδιαγραφές. Σας ερωτώ λοιπόν, ως πρόεδρος της COP21, τι μπορεί να γίνει ώστε αυτή το, η συνολική προσέγγιση εμπορίας ε, λοιπόν να συνδυαστεί με αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ. παρακαλώ. Τους μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας πρώτα απ' όλα και καλώς ήρθατε. Είσαστε εσείς ο αμφιτρίωνας της COP21 στο Παρίσι. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι δυνατόν στο τέλος σε σχέση με τη σύνταξη του εγγράφου για τα συμπεράσματα το σχέδιο το προκατακτικό για τη διάσκεψη αυτή όπου ο τομέας των μεταφορών, εναέριων μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών δεν εντάσσεται Δηλαδή κάνουμε λόγο για τις διεθνείς οργανώσεις ε, εναέριας με εναέριων μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος, κάνετε λόγο για τόσες πολλές παρεμβάσεις από όλες τις χώρες, πράγμα μεγάλης σημασίας. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει στο να καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Όμως πώς είναι δυνατόν να φτάσουμε στο τέλος χωρίς να υπάρχει δέσμευση, αν μπορώ να το πω έτσι, αν αυτές οι οργανώσεις εναέριων μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών δεν εντάσσουν στο έγγραφο. Ευχαριστώ. Now... ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που προσήλθατε σε μας. Μια απλή ερώτηση. Πριν από δύο εβδομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων ψηφίσαμε, υπεψηφίσαμε μια δική μου τροπολογία λομπιστική δραστηριότητα όπως και στη διάσκεψη των Παρισίων ε, ε, διαφαίνεται θα πρέπει η ημερήσια διάταξη της COP21 να μπορέσει να διαμορφωθεί με ένα ανοιχτό τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμη για όλους όσους ενδιαφέροντα συμμετάσχουν. Η επιτυχία της διάσκεψης ε, θα έχει τεράστια σπουδαιότητα. Εδώ εκείνοι που έχουν περισσότερη εξουσία από τους πολίτες και χρήματα και εκπροσωπούν πολύ σημαντικά συμφέροντα. Είσαστε εσείς πρόθυμος να δεχτείτε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ίση πρόσβαση και όλες οι, δια, διαστηριότητες των λομπιστών πρέπει να είναι διαφανείς. Συμφωνείτε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Υπουργέ που είστε παρόν. Να αναφερθώ στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε μία-δύο φορές η χρηματοδότηση, δεν θα το επαναλάβω αυτό. Αναφέρομαι στην περίοδο δέσμευση για την πενταετία. Στις διπραγματεύσεις όλο και περισσότερες χώρες δεσμεύονται για πενταετία. Και είπατε πόσο χρήσιμο, πόσο κρίσιμο ήταν να μην έχουμε πολύ μακροσκελή περίοδο για την οποία δεσμευόμαστε. Έχει τεράστια προβλήματα η Ευρώπη, διότι έχουμε ένα στόχο για το 2030 και τίποτα για το 2025. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα και ίσως μια συμβουλή να σας δώσω. Πώς μπορούμε να πάμε προς το στόχο του 2025. Έφυγε ο συνάδελφος του UKIP, ο κ. Χέλμερ, που πάντα ισχυρίζεται ότι όλοι φεύγουν από την Ευρώπη λόγω της ε, πολιτικής για το κλίμα. Ε, είναι επίκαιρο λοιπόν το θέμα. Θέλω να πω λοιπόν, διαβάστε τις ε, διάφορες εκθέσεις. Μείον 23% καταφέραμε μείωση. Έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας. Οποιαδήποτε μηχανία κλείνει δεν είναι λόγω της πολιτικής για το κλίμα. Το μείον 40% το στόχο μπορούμε να τον κάνουμε στόχο για το 2025. Θα είναι καλό αυτό αν γίνει στο Παρίσι, θα μας βοηθήσει όλους και θα είναι ένα καλό μήνυμα που θα αφορά την αξιοπιστία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη αυτή τη συμβουλή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών. Μας είπατε σήμερα ότι τρεις παραμέτρους ε, θεωρείτε ότι είναι ε, σημαντικές ε, για την επιτυχία του COP21. Δεσμευτικές πρέπει να είναι οι ε, διατάξεις αυτές νομικά. Μπορούμε να σας συγχαρούμε. 90% έχουν κατατεθεί οι προτάσεις. 154 χώρες σε σχέση με το Κιώτο είναι πολύ φιλόδοξο και ο στόχος των δύο βαθμών Κελσίου δείχνει ότι είναι και λογικό το πλαίσιο. Δεσμευτικά όλα από πλευράς νομικών. Ε, μεγάλη πρόκληση για τις 154 χώρες που δεν κατάφεραν να, να δεχθούν αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα. Στην Κίνα, όταν θα έχετε επαφές με την κινέζικη κυβέρνηση, να τους πείτε ότι χρειάζεται αυτός ο δεσμευτικός χαρακτήρας. Οι μεγαλύτερες εκπομπές τρύπων από τις αναδυόμενες χώρες ε, προέρχονται και το burden sharing μεταξύ φτωχών και πλουσίων είναι σημαντική υπόθεση ο επιμερισμός ευθυνών. Και για το Ταμείο μέχρι το 2020 καλή πρόταση αυτή. Ωστόσο Μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει ένας ε, φόρος, ε, ένα τέλος συναλλαγής ε, επί των χρηματοοικονομικών πράξεων. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα αυτό. Τι βρίσκεται επί τραπέζης ακριβώς. Συνάδελφοι, έχουμε 27 συναδέλφους να μιλήσουν. Σας παρακαλώ. Χάιντς Φλόρεντς. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιάστηκα Μικρόφωνο να μιλάει πιο καθαρά ο μιλητής. Μάλιστα ήμουνα και κάτω παρελθόν παρόν και μπορώ να σας πω ότι η γαλλική δημοκρατία είναι πολύ σημαντική στην διάσκεψη των Παρισίων με την παρουσία της. Εμείς ε, εσείς ε, μπορείτε να εγγυηθείτε αυτή την επιτυχία ε, κανείς άλλος και να μην είμαστε υπερβολικοί στο εγχείρημά μας. Μετά θα ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι. Το καλύτερο παράδειγμα ήταν το Μεξικό. Θετικό αυτό και υπήρξε και στο βορρά της Ευρώπης ε, μια ε, αρνητική εξέλιξη. Είναι στα χέρια σας ε, και των συμμάχων σας και των Υπουργών Εξωτερικών στις επαφές σας να προχωρήσετε. Αφήστε τους απεσιόδοξους στο σπίτι τους, στις χώρες τους και μην συνασπιστείτε με τους ακραίους πρασίνους, με τους λογικούς να απορρευθείτε και θα βοηθήσει αυτό περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ο κ. Γραμματικάκης. Το μικρόφωνο σας. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εισήγηση του κυρίου Υπουργού, πράγμα που συμβαίνει σπάνια στις αίθουσες του Κοινοβουλίου, γιατί είχε λιτότητα, δηλαδή ήταν σύντομος και επίσης μίλησε ουσιαστικά. Ε, επειδή εγώ κύριε Υπουργέ είμαι ένας καθηγητής φυσικής θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο με σας και να σας πω ότι ο στόχος του 2,7 βαθμών που θέσατε είναι μεν αισιόδοξο, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι αρκετός γιατί τα νέα δεδομένα ίσως το ξέρετε αλλά και τα ορατά κλιματικά φαινόμενα έχουν δώσει μια εικόνα του πλανήτη στο έλεος, στο χείλος του γκρεμού Βέβαια καλό θα είναι και τα δύο ή τα τρία ή τρεις βαθμοί μέσα στις ε, συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά υπάρχει μία ιδέα που κυκλοφορεί πολύ καιρό τώρα. Δεν πήρα όμως απάντηση. Μήπως δηλαδή μία λύση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να είναι οι δημόσιες επενδύσεις που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ελάχιστε σε όλες τις χώρες και να έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και στις χώρες που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία να υπολογίζονται στον υπολογισμό των ελλημάτων. Αυτό φυσικά έχει πολλά πολιτικά εμπόδια, αλλά η ικανότητά σας μπορεί να τα ξεπεράσει νομίζω. Η ιδέα των ελικοπτέρων που θα παρακολουθούν λίγο την κλιματική αλλαγή μου άρεσε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι από τον, στον Άρη ανακαλύψαμε νερό. Πολύ εύκολο θα δούμε τη ρήπανση στα κράτη. Τη φοβάμαι όμως λίγο. Έχουν παραγίνει κατασκοπευτικοί δορυφόροι. Ελπίζω ένας, να μην είναι ένας από αυτούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. And now, Ms. Κυρία Βιτσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζουμε τώρα σε σχέση με τις δεσμεύσεις ε, που έχουν αναλυθεί για αυτή τη διάσκεψη των Παρισίων. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις αυτές είναι διαφορετικές μεταξύ τους και είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους γίνεται λόγο για διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού και κάποιοι από τους ε, μεγαλύτερους ε, από πλευράς εμπλοκής ε, δεν δεσμεύονται καν σε σχέση με τις εκπομπή Αυτό το χάος λοιπόν μπορεί να είναι σχεμένο ε, για να αποφευθούν κοινά συμπεράσματα και δεσμεύσεις ε, σε σχέση με την ε, εμπλοκή και την υπογραφή από όλους μιας τέτοια συμφωνίας όπως αναφέρατε σημαντικό αυτό όμως θα έπρεπε από την άλλη πλευρά να κάνουμε λόγο και για άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε. Ευχαριστώ Υπουργέ. Συμφωνούμε όλοι ότι η διάσκεψη κορυφή των Παρισίων πρέπει να στεφθεί με πτυχία και με, συγκαταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών κτλ. Αυτό που με ανησυχεί είναι μετά από την ε, γνώση μα των δηλώσεων σε σχέση με το τι συμβαίνει από πλευρά ε, Ηνωμένων Πολιτειών ε, και ε, δεν ξέρω το τι πρέπει να γίνει. Σα ερωτώ, πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δυνατότητα να μειωθεί η αύξηση της θερμοκρασία ε, κατά δύο βαθμού όταν χώρε όπω η Κίνα για παράδειγμα δεν είναι πρόθυμες να καταβάλουν καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ και ο Τζάμπορ. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ που είστε εδώ μαζί μας. Έχω μια ερώτηση, μόνο μια ερώτηση συγκεκριμένη. Αναφερθήκατε εκτενώς στην θέση του Κοινοβουλίου ε, την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου που υιοθέτησε επίσης μια αναψήφισμα που αφορούσε τους, ε, την νομοθεσία για το κλίμα. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα που πετύχαμε θα βγουν εκτός του TTIP και το ISDS. Δηλαδή το μηχανισμό διευθετήσεως των διαφορών. Θα βγουν εκτός της δικαιοδοσίας αυτών των εργαλείων, ούτως ώστε να μην υπονομεύσουμε τα επιτεύγματα όσον αφορά το κλίμα, αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε να τα θυσιάσουμε στο βωμό των οικονομικών ε, κερδών. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν έχει συγκεκριμένη θέση από αυτού. Διερωτώ η φιλοξενούσα χώρα την οποία εκπροσωπείται αν η Γαλλία θα υποστηρίζει τη θέση μας αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ είμαι, καλημέρα. Μπορώ να είμαι πολύ λακωνικό. έχω την ίδια ερώτηση ο κύριο Γκρέτε και ο κ. Ντάνκαν όσον αφορά το ETS, το σύστημα ανταλλαγή των ε, ρήπων, εμπορία ρήπων. Διότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία θα ήταν να συνδέσουμε το σύστημα αυτό με άλλα συστήματα παρόμοια στον κόσμο, σε άλλα μέρη του κόσμου. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού, διότι όπως και η κυρία Γκέρλινγκ είπε, θα αποτελούσε απάντηση στις ανάγκες της βιομηχανίας, στη χαλιβουργία, παραγωγή τσιμέντου κλπ. που αντιμετωπίζουν ε, αθέμητο ανταγωνισμό. Ποιε είναι οι προοπτικέ στο Παρίσι λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα σύστημα παγκόσμιο εμπορίου λοιπόν, παγκόσμιο ETS. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπράνον. Ευχαριστώ Υπουργέ. Δύο ερωτήσεις. Το ευρωπαϊκό κοινό γνωρίζει όλο και περισσότερο τι ρόλο παίζουν τα ρηκτά καύσιμα στην αλλαγή του κλίματος δεν γνωρίζουν όμως τόσο πολύ το ρόλο που παίζει η γεωργία στην αλλαγή του κλίματος. Συμφωνείτε ότι η γεωργία θα πρέπει να υπομειστεί το βάρος που της ανήκει στην αντιμετώπιση αλλαγής του κλίματος και ότι η γεωργία δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Όλοι γνωρίζουμε καλά το, το κόστος για το περιβάλλον που έχει το κοινοβούλιο που έχει δύο έδρες και σαν ε, θέλω μια συμβολική πράξη γαλλική. Αν η γαλλική κυβέρνηση μπορούσε να υποστηρίξει μία έδρα για το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένη που είστε εδώ κύριε Υπουργέ για να συζητήσετε μαζί μας τα επίπεδα της Επιτροπής Περιβάλλοντος το θέμα αυτό. Έχω μια ανησυχία όσον αφορά την ομάδα G77 που έχει πάνω από 134 χώρες ε, Νότια Αφρική, Κίνα κλπ. μεταξύ αυτών. Σαν συμπρόεδρος λοιπόν των χωρών ΑΚΕ, ε, των επαφών με τις, τις με τις χώρες ΑΚΕ, ε, βλέπω ότι έχουν μεγάλη καχυποψία ενώ των επιτυγμένων χωρών οι ανεξόμενες χώρες τα 62 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο ΣΑΙ τη είπαν αντιστοιχεί σε εμά. Δεν μα επέτρεψε σε εμά να προσαρμοστούμε όσον αφορά την άνθιξη τη θερμοκρασία. Εξού και το πολύ διπλωματικό μου ερώτημα, και ξέρετε ότι παίζεται ρόλο σε αυτό. Πώ λοιπόν, τι μπορούμε να συζητήσουμε με τι χώρε αναπτυσσόμενε. για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Ευχαριστώ κυρία Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. 126 χώρες από 155 έχουν υποβάλει τη συνεισφορά τους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός από τη ΣΥΠΑ, η κάθε χώρα το έχει κάνει με διαφορετικό τρόπο και με βάση διαφορετικές πολιτικές. Δεν θα πρέπει να εναρμονιστούν όλα αυτά κατά τη γνώμη σας. Ιδαλλιώς τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα δεν θα είναι ποτέ αξιόπιστα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικός ο μηχανισμός εποπτείας, παρακολούθησης, επαλήθευσης και κοινοποίησης, γνωστοποίησης. Η Επιτροπή είπε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε διεθνείς εμπειρογνώμονες που θα τα ελέγχουν όλα αυτά αλλά οι περισσότερες χώρες πιστεύουν ότι είναι παρέμβαση στα εσωτερικά τους πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα γιατί αυτό που είναι αναγκαίο είναι πραγματικά αναγκαίο έτσι δεν είναι ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ Υπουργέ που έρχεστε να μας μιλήσετε. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ερώτηση έχω. Θέλω δύο οπτικές γωνίες επ' αυτού. Ποια είναι η άποψή σας για την Ενεργειακή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, Ενεργειακή Ένωση, πώς τη βλέπετε σαν εργαλείο που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τα συνέπειες αλλαγής του κλίματος και να πετύχουμε τους στόχους του COP21. Δεύτερη οπτική γωνία, Ενεργειακή Ένωση, σαν εργαλείο που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τους ισχυρισμού κάποιων επιθετικών χωρών όπως η Ρωσία που προσπαθούν να επηρεάσουν την εξωτερική μας πολιτική. Τις αξιώσεις τους μάλλον. Ο κ. Σαφχάουζα. Κύριε Υπουργέ, όταν ήμουν επικεφαλής της Επιτροπής Ενέργειας, ο Κλοντ Ζιρόν μου έλεγε ότι δεν θα κάνεις τίποτε αν δεν υπάρχει πολιτική τιμών όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Σήμερα η τιμή των, των ορυκτών καυσίμων μειώθηκε πάρα πολύ. Άρα, πρώτη ερώτηση. Μπορούμε μήπως να επηρεάσουμε αυτούς που ξέρετε το κατάρτι, τη Σαουδική Αραβία, όλους ιδιαιτέρως ούτως ώστε να αλλάξουν την πολιτική τιμολόγηση. Και αν θέλουμε να επιταχυνθεί η διαδικασία πρέπει να αυξηθεί η τιμή των ορυκτών καυσίμων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Την χειραγωγούν αυτή την τιμή. Από πλεόνασμα τεχνητό ή έλλειψη τεχνητή των ορυκτών καυσίμων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση. Είναι θεμελιώδου σημασία αυτό τη επενδύσει, να σταθεροποιηθεί η τιμή. Μια σταθεροποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επενδύσει μέσω μηχανισμού σταθεροποίηση για τι νέε τεχνολογίε. Μετά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, είναι η ποσοτικοποίηση ε, χρειάζεται ένα τρισεκατομμύριο στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης. Ελάχιστον αυτό. Λοιπόν, ε, γιατί να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ποσοτικοποίηση για την ενεργειακή μετάβαση. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δύο σύντομε ερωτήσει αν επιτρέπετε. Εγώ ίδια ήμουν εισηγήτρια για τη συντάκτη γνωμοδότηση Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτό το ζήτημα. Και το ερώτημα είναι πώς θα το καταφέρετε οι διαπραγματεύσεις TTIP για τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματα της COP21 για την προστασία του κλίματος και δεύτερον για την κλιματική διπλωματία. Σύντομα αναφερθήκατε εσείς σε αυτό το θέμα. Είπατε ότι στις 10 Νοεμβρίου θα συνέλθετε εκ νέου. Ερώτηση όμως, πώς η κλιματική διπλωματία μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσει ώστε οι χώρες που πλήττονται με ιδιαίτερο τρόπο από τις κλιματικές αλλαγές να ενταχθούν περισσότερο σε αυτόν τον κύκλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είμαι συγγετής για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Με ενδιέφερε αυτό που είπατε για δεσμευτική συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς θα επιβληθεί όμως μετά από πέντε χρόνια. Τι θα χρησιμοποιήσουν τακτική να πούμε ότι αν όλες οι χώρες ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους ίσως αναθεωρήσουμε προς τα πάνω το στόχο για το 2030 και αν όχι θα αναθεωρήσουμε προς τα κάτω το στόχο. Κυρίως αν τα στοιχεία οδηγούν να δείχνουν ότι υπάρχει διαρροή άνθρακος, όπως ανέφεραν προελίσσατες, για τη Γεωργία. Με την πράσινη της ΚΑΠ έγινε πολύ πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον η Γεωργία. Υπάρχει και ένας φόβος. Αν δεν αναγνωριστεί η σύλληψη του άνθρακα και αποθήκευση του άνθρακα χάσει στη Γεωργία θα έχουμε ξανά διαρροή άνθρακα που θα είναι πιο επιβλαβής για το περιβάλλον το ερώτημα του κυρίου Λίζε για την αυσιπλοεία και την αερο, τις αερομεταφορές. Έχω και εγώ την ίδια πορεία. Τέλος, εξίσου, σημαντικός ο κύριος Πέτερλε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα αν βάλουμε τους φιλόδοξους στόχους σε ευρύ πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάσουμε τους κλιματολογικούς στόχους με τους αναπτυξιακούς στόχους των εταίρων μας. Η Ινδία είναι ένας από τους σημαντικότατους εταίρους που προβλέπει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την επόμενη 20 ετία. Συνέπεια θα είναι τριπλάσια εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακος αν ακολουθηθεί το κινέζικο μοντέλο. Χρειάζεται στρατηγική αλλαγή όσον αφορά τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ινδία θα πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να συμμετάσχουμε στο να γίνει πιο οικολογική η ειδική οικονομία. Είναι εφικτό. Ερώτηση κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε αυτή την πρόκληση. Τι δέσμευση θα αναλάβετε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας εύχομαι μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι και μετά τη διάσκεψη. Επίσης, ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση, ο κύριος Τούρμες. Κύριε Υπουργέ, μου λένε ότι κάντε με καλό ντουέτου με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και χαίρομαι πολύ. Ε, πρέπει να προσανατολιστώ επί των λύσεων. Και μία από τις λύσεις είναι να πηγές ενέργειας. Ένα ελάχιστα γνωστό ε, πρόβλημα γιατί έχει περισσότερο, χρησιμοποιείται περισσότερο ηλιακή ενέργεια στην ε, ε, Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Υπάρχει, περισσότερο ήλιο στην Ελλάδα, αλλά το κόστο το το του κεφαλαίου, το spread, ε, το διαφορά κεφαλαίου μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία είναι περισσότερο από τη διαφορά του ηλίου. Το ίδιο και για την Αίγυπτο και τι αφρικανικές χώρε. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να λυθεί για να χειριστούμε τι επενδύσει είναι πρέπει να βρείτε στο Παρίσι έναν μηχανισμό ένα, ένα ταμείο που μειώσει του κινδύνου, να εμποδίζει αυτό το φαινόμενο, να, να μειωθεί το κόστος του κεφαλαίου, να είναι πιο χαμηλό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις χώρες εκείνες που ε, τιμωρούνται από τις σηματοστικές αγορές. Στην Αίγυπτο πληρώνουν 20% το ΟΚΟ, 4% στη Γαλλία, 2% στη Γερμανία. Ε, αυτό είναι σημαντικότατο εργαλείο. Τελευταίο ε, παράδειγμα, ε, μάλλον ερώτημα. Το Nord Stream είναι ένα θέμα που διχάζει την Ευρώπη. Η Gaz ε, de France κλπ. Ίσως θα, έπρεπε να, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί, να επανεξετάσει τη θέση της η Ευρώπη πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαμπιούς, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ δύσκολο να απαντήσω σε 10 λεπτά, αλλά 10 λεπτά έχω στη διάθεσή μου. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματά σας πράγματι. Παρόλα αυτά ε, χρειαστήκατε σχεδόν μισή ώρα για να τα θέσετε. Αυτή είναι η ελευθερία κοινοβουλευτική. Επομένως μην μου κρατήσετε κακία αν δεν μπορέσω εγώ να απαντήσω μέσα στα 10 λεπτά. Να σας πω ότι έχω σημειώσει. Καταρχάς, υπήρξαν ερωτήσεις για τον ε, τομέα των θαλάσσιων και αέριων μεταφορών. Σας παραπέμπω στο κείμενο της Βόνης που εγκρίθηκε στη Βόνη την περασμένη εβδομάδα. Το άρθρο 3 στο εδάφιο 17 ε, ασχολείται με αυτό το θέμα με μια σύντομη διατύπωση το δέχομαι και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό θα πρέπει το θέμα να το συμπεριλάβουμε στον ευρύτερο προβληματισμό μας, γιατί είναι σημαντικός. Όμως σας παραπέμπω στο άρθρο 3,17. Πολλοί εξ ημών αναφέρθηκαν στη, στο κόστος του άνθρακα και στη τιμή του άνθρακα. Και αν ε, η Κίνα ε, θα ε, συμβάλλει στη σωστή κατεύθυνση. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη για τον άνθρακα. Είναι απαραίτητο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλες οι αποφάσεις δημοσίων χρηματοδοτήσεων που παίρνουμε ως αποφάσεις και που είναι απαραίτητες είναι δεν είναι τόσο σημαντικές λόγω του μεγέθους τους, αλλά είναι σημαντικές γιατί μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλό στο μηχανισμό της αγοράς και να επιφέρουν εκεί ε, ε, μεταγενέστερα ε, μεγάλες αλλαγές. Αν έχουμε ε, τιμολόγηση του άνθρακα, και σημειώνω αυτό που λέτε για τα, για του ήλιου. Έτσι τροποποιούμε το πώς θα τοποθετηθεί η αγορά. Όλο το σύστημα το αλλάζουμε και γι' αυτό πρέπει προς τα εκεί να κινηθούμε. Σήμερα το πρωί στο κινητό μου διάβασα για μια συνάντηση που έγινε στην Ινδία. Πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω αν την έχετε μάθει. Μια χώρα πληθυσμού 1,5 δις κατοίκων μου είπε διαμέσου του Προέδρου της ότι και ας πούμε στη θέση της θέλω να συμβάλλω μου είπε ο Πρόεδρος της χώρας αυτής αλλά έχω 500 εκατομμύρια ανθρώπους που πρέπει να βγάλω από το όριο της πτώχειας και το, η μόνη πηγή ενέργειας που έχω είναι ο άνθρακας βοηθήστε με μου είπε λοιπόν να πάω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σιγά σιγά. Και η χώρα αυτή με άλλες χώρες θα συνάψει συμμαχίες για την ε, ηλιακή ενέργεια και θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι έτσι ώστε να ε, ανταποκριθούν στα δέοντα. Ξέρετε, ως προς την Κίνα θα πάμε στα τέλη αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επομένης. Θα έχουμε κοινή δήλωση και σε αυτή τη δήλωση έχουμε προβλέψει να γίνει αναφορά στην απόφαση των Κινέζων για το 2017. Οπότε και θα ε, ε, συστήσουν αγορά άνθρακα με τιμή. Κειμενόμενοι εκεί. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η τιμή του άνθρακα είναι χ για όλο τον κόσμο συγκεκριμένη. Όμως βλέπουμε παντού πρωτοβουλίες που συγκλίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και υπάρχει και μια έκθεση που εξετάζει τις διάφορες τεχνικές και μιλά για έναν ενεργειακό διάδρομο του άνθρακα ως προς την τιμολόγησή του. Πολλά και διαφορετικά στοιχεία συγκλίνουν σιγά σιγά. Ελπίζω ότι Συμφωνία των Παρισίων θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι στην συγκεκριμένη χώρα π.χ τη Γουατεμάλα ε, θα μπορούμε να πούμε ότι η τιμή του άνθρακα θα είναι τόση δεν έχουμε αυτή την εντολή ούτε αυτό το δικαίωμα ελπίζω όμως ότι στη διάσκεψη των Παρισίων ε, θα βλέπουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να συγκλίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και τελικά η δημόσια παρέμβαση θα λειτουργήσει ως μοχλός που θα κινητοποιήσει την αγορά και θα αλλάξει το σύστημα από εκεί και πέρα ως προς τις επαληθεύσεις Πράγματι είναι ετερογενείς οι συνεισφορές της κάθε χώρας μέλους, του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλλει δηλαδή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πέρσι στη Λίμα μπορέσαμε να φτάσουμε σε συμφωνία μόνο δεχόμενοι ότι για πρώτη φορά η συνεισφορά της κάθε χώρας να είναι έστω ετερογενής. Αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει σε συμφωνία Είναι μόνο αυτές οι διατάξεις που μπορούσαμε να δεχθούμε. Δεν μπορούσαμε να έχουμε συγκεκριμένες πολύ αυστηρές προδιαγραφές γιατί οι χώρες δεν θα τις δέχονταν. Δεχτήκαμε δηλαδή την ετερογένεια προκειμένου να ε, συμβάλλουν οι χώρες. Ορισμένες από αυτές τις συνεισφορές είναι απόλυτες και άλλες είναι υποαίρεση κυρίως ε, των ε, φτωχών χωρών μελών. Λέει μια χώρα αυτά δεσμεύομαι να κάνω ούτως ή άλλως και δεσμεύομαι να κάνω και άλλα τόσα εάν μου δώσετε τεχνολογία και δυνατότητες και μέσα. Ε, για λόγους ρεαλισμού ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό. Μου τέθηκε μια ερώτηση για τη διαφάνεια, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπά. Δεν γνωρίζω τι διαβουλεύσεις είχατε εσείς, αλλά το θέμα τίθεται ούτως ή άλλως. Στην ε, σύσκεψη της Βόνης ελήφθη η απόφαση με βάση την πρόταση της Ιαπωνίας, όχι για τα λόμπι αλλά για τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να πούμε δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε ε, πολλά πράγματα, μπορούμε να διαπραγματευτούμε με πλήρη διαφάνεια και σε άλλους τομείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε παρουσία των διαπραγματευτών. Δεν είναι και το πιο εύκολο να ε, γίνει, πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί, έναντι των παρατηρητών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από την άλλη πρέπει να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και γνωρίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια ότι εάν όλα είναι ανοιχτά, ανοιχτή προσέλευση σε όλες τις συζητήσεις ε, θα έχουμε 20.000 αντιπροσώπους και 5.000 ε, δημοσιογράφους ε, σε μία σύσκεψη. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι. Δεν αναφέρομαι τώρα στα λόμπι είναι μια δύσκολη ε, διοργάνωση και τεχνικά μελώντας. Βεβαίως ε, έχουμε κάνει τα πάντα έτσι ώστε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να είναι παρούσες και να τιμούμε την έννοια της σύγχρονης δημοκρατίας. Τώρα, η ομάδα των 134 χωρών είναι αρκετά επιφυλακτική ε, ως προς τις πλούσιες χώρες και καλούμαστε εμείς να υπερπηδήσουμε αυτήν την τροχοπέδη, να δείξουμε ότι δεν έχουμε κρυμμένη πολιτική ατζέντα και θα πρέπει και οι χώρες αυτές <clears throat> να καταλάβουν ότι έχουν υπάρξει διάφορες εξελίξεις γιατί αν δούμε τον κατάλογο των πλούσιων χωρών και τον κατάλογο των μη πλούσιων χωρών που, είχε, ε, που είχαν συνταχθεί πριν από 25 χρόνια και δούμε και τη σημερινή κατάσταση ε, έχουν φύγει αντιστοίχω από τον μεν και τον δε. Ε, κάποιες αναδυόμενες χώρες έχουν πλέον αναδυθεί. Θα πρέπει να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, τα μέτρα που θα πάρουμε για την προσαρμογή στην έκθεση του ΟΣΑ, το ενδιαφέρον και το ανδιαφυσβήτητο είναι ότι υπάρχει χρηματοδότηση σημαντική για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά όχι επαρκής χρηματοδότηση για την προσαρμογή. Το σύνολο που έχει δοθεί είναι συγκεκριμένο και 16% του συνόλου αυτού μπαίνει στην, και κατευθύνεται στην προσαρμογή. Παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν την σημασία του μετριασμού του φαινομένου, η προσαρμογή είναι το πιο σημαντικό γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε αποτελέσματα και τώρα και μετά από 25 χρόνια. Και μάλιστα πριν από το 2020 θα πρέπει να επιτευχθούν πολλά από αυτά. Η Συμφωνία των Παρισίων θα αρχίσει να ισχύει ε, το 2020. Αλλά πέντε χρόνια μεσολαβούν μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Υπάρχει μια πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία Cruise ε, είναι τα αρχικά για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όλων των ενδιαφερομένων ατόμων από την έλευση και εμφάνιση καταστροφών, φυσικών καταστροφών. Υπάρχει ένα σύστημα αντασφάλισης το οποίο μελετά τώρα η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Αφρικής. Ξέρετε, μόνο το 25% της 100 της, Αφρικής, ε, της Αφρικανικής Υπήρου έχει ηλεκτρισμό και υπάρχουν ε, τρόποι για να αλλάξει πραγματικά η ζωή του κόσμου εκεί. Έχω φίλους στην κυβέρνηση του Μπενίν που έχουν ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο στοιχίζει μόνο κάποιες δεκάδες ε, εκατομμύρια και που θα επιτρέψει να υπάρξει σύνδεση του μισού πληθυσμού. Και άρα τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν τα μαθήματά τους το βράδυ. Ενώ τώρα υποκείται μόνο ε, στο, ε, εξαρτώνται μόνο από το πότε έχει φως από τον ήλιο. Άλλωστε, πολύ συχνά είναι ο μόνος τρόπος να εμποδίσει κανείς ε, τα ε, φίδια να μπουν μέσα στις καλύβες ή αλλού. Βλέπετε ότι έχουν ένα σχέδιο στο Μπενίν που στοιχίζει μόνο λίγες δεκάδες εκατομμύρια ε, ευρώ ή δολάρια και μπορεί να δώσει ρεύμα στο μισό πληθυσμό με τεράστιες θετικές συνέπειες, με τεράστιο θετικό αντίκτυπο. Σε κάθε περίπτωση Η Γαλλία είχε πάρει την πρωτοβουλία για, την, για το 4 επί 1000 ε, και άλλες χώρες, ούτως ώστε να υπάρξει ε, χρηματοδότηση του Ταμείου και κεφαλαιοποίηση αυτού. Πολλοί από εσά είπατε ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το Στρασβούργο ως έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λόγους περιβαλλοντικούς. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πραγματικότητα. Υπάρχουν, υπάρχει κείμενη νομοθεσία επ' αυτού. Άλλωστε, αν ήταν το περιβαλλοντικό ε, κριτήριο ε, το μόνο, ε, τότε να επιβάλλουμε σε όσους πρέπει να πάνε στις Βρυξέλλες, από όπου και αν προέρχονται, να πάνε με το ποδήλατο. Άλλωστε, υπάρχουν και άλλες διατάξεις που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Κλείνοντας, ε, ε, ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήμουν εξαιρετικά σύντομο στις απαντήσεις μου, αλλά αν ήμουν πιο μακροσκελής θα είχα πάρει πολύ από το χρόνο σας. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι είναι μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας. Η Γαλλία είναι η χώρα οικοδεσπότης. Να μην το συγχαίουμε. Το συγχαίουμε. με τον Παντοκράτορα. Άλλο οικοδεσπότης, άλλο Παντοκράτορας. Θέλω όμως να αναφερθώ στο Περού που υποδέχτηκε τη διάσκεψη πέρσι. Ε, και η χώρα αυτή έκανε μια πολύ καλή δουλειά και φέτος έχουμε δουλέψει πολύ με τους φίλους μας από το Περού. Το Περού είναι μια ε, χώρα φτωχή υποτίθεται του Νότου και συνεργάζεται με μια χώρα όπως τη Γαλλία του Βορρά και πιο ε, πλούσια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει ένα μήνυμα ελπίδας και εμπιστοσύνης και στους μεν και στους δε. Να είστε σίγουροι ότι με τη δική σας στήριξη θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε. Η Ευρώπη σε αυτή την υπόθεση έχει ρόλο κλειδί να διαδραματίσει. Μπορεί κανείς να πει ότι όντως η Ευρώπη να είναι ανεπαρκή στο χύψη σημείο. Επιμέρους, τμηματικά, ωστόσο, είναι η μία από τις υπήρους, για να μην πω η μόνη, που πραγματικά δείχνει το δρόμο. Δείχνει leadership, πάλι εισάπτες στον γαλλική θα το πω. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικά ε, τα βήματα της Ευρώπης όχι για να επιβάλλει οτιδήποτε άλλωστε νομικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στον οποιοδήποτε οτιδήποτε αλλά για να δείξει η Ευρώπη ότι είναι δεσμευμένη προς μια αλλαγή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί να συνεχίσει να είναι βιώσιμος ο πλανήτης μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εδώ ολοκληρώνατε η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Να επενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. We received useful information.